με ομοφωνία. Όλα τα παραδείγματα που σας έδωσα, όλα αυτά τα πέντε ζητήματα είναι μπλοκαρισμένα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σας κάνω λοιπόν έκκληση τώρα και στα επόμενα χρόνια να δώσετε αυτή την πολιτική μάχη που πρέπει να δώσουμε γιατί διαφορετικά θα μείνουμε σε ευχολόγια που ποτέ δεν θα υλοποιηθούν. Και κύριε Πρόεδρε, πρώτη φορά έκανα κάτι αδύνατον μόλις έμεινα στα τέσσερα λεπτά μου κύριε Πρόεδρε. Ναι, η κυρία Κέλλερ για τους ε, πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας. Πιστεύω ήταν πολύ φιλοευρωπαϊκή και ισχυρή και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί πολλοί ανησυχούν όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, πολλές ε, κυβερνήσεις ε, αποτυγχάνουν στην εξασφάλιση του κράτους δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα τη. Άρα είναι θετικό το ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε τα πράγματα μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Αυτό είναι πολύ καλό. Και θα ήθελα να συγχαρώ επίσης για όλα τα μέτρα τα οποία λήφθησαν στην Ισπανία και που αντανακλούν ακριβώ τι δεσμεύσει που εξφράσατε εδώ και την απόφαση σα, για παράδειγμα, να αυξήσετε τον ελάχιστο μισθό ε, των 900 ε, ευρώ. Κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλέ οικογένειε. Επίση, συνδυασμό με με, τις, με, με τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος που είναι μια μεγάλη βελτίωση. Εμείς επιθυμούμε μια κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες στο Συμβούλιο και στις χώρες μέλη και ελπίζω και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Και δεύτερον η απόφασή να εξασφαλίσετε ε, η, τα νοικοκυριά να βάλουν ε, ε ηλιακό, ηλιακές εγκαταστάσεις στην, ε, στις στέγες τους. Ε, ε ούτως ώστε ο καθένας ε, μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη. Χρειαζόμαστε αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, ε, χάρηκα, γιατί όπως επαναφέρατε, η κυβέρνησή σας έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και απέχουμε πάρα πολύ από μια ε, δρέωση τη ισότητα των φίλων. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες γιατί Υπάρχουν ε, πολλέ χώρε που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών και είναι πολύ θετικό να υπάρχουν κυβερνήσει που προωθούν μια φιλόδοξη ε, ατζέντα που είναι υπέρ τη ισότητα των φύλων. Βεβαίω το έργο είναι δυσχερέ, κληρονομήστε πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η κατάσταση στην Καταλωνία. Ε, και, και ο προκάτοχός σας υπήρξε εξαιρετικά αδιάλακτος. Τώρα έχετε εσεί το θέμα στο τραπέζι σας και είναι ξεκάθαρο ότι μόνο μια δημοκρατική πολιτική λύση θα μπορούσε να οδηγήσει την Ισπανία μπροστά και περιλαμβάνει επίση μια λύση και για τους φυλακισμένους, επίσης τα πρώην μέλη τη δική μα πολιτικής ομάδας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις φυλακές. Ε, ε, χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος γιατί μόνο με μια θετική βούληση και από τις δύο πλευρές ε, θα έχουμε αποτελέσματα και θα έρθουμε πιο κοντά σε μια λύση που χρειάζεται κατεπηγόντως για την Καταλωνία, για το σύνολο της Ισπανίας και για ολόκληρη την Ευρώπη. Αναφέρεται κύριε Πρωθυπουργέ τις ευρωπαϊκές αξίες και εδώ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όταν βλέπουμε την κατάσταση στην Ανδαλουσία και το σχηματισμό της τοπικής κυβέρνησης εκεί. Γιατί ένα ακροδεξιό εξερμιστικό κόμμα θα συμπεριληφθεί στην κυβέρνηση. Γίνεται ανεκτό και λυπούμε που η συντηρητική και οι δεξί συμφωνούν ε, γι' αυτό. Ε, και ε, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτά συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες και δεν χαίρονται για αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλυφθεί συγκεκριμένη δράση. Όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να προσπαθήσουν να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά είναι επονίδιστη συμφωνία όταν μια πολιτική ομάδα δέχεται να συνεργαστεί με ένα ακροδεξιό κόμμα. Εμείς ε, υποστηρίζουμε τις γυναίκες που αυτή τη στιγμή δηλώνουν για την ισότητα των φύλων, γιατί η βία κατά των γυναικών δεν έχει καμία θέση οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι πολλοί από τους στόχους που αναφέρατε, ισότητα των φύλων, κοινωνική Ευρώπη κλπ. Όλα αυτά προποθέτουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν ελπίζουμε ε, τις δικές σας πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο, να ε, στηρίξετε το Συμβούλιο σε αυτή την κατεύθυνση και να εξασφαλίσετε οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο επίσης να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση μιας σοσιαλιστικής και φιλοδημοκρατικής ε, Ευρώπης. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ΓΟΥΗ, κυρία Λόπες Βερμέχου. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τσάντσε, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ παρόν και για το ότι συμβάλλεται στην ευρωπαϊκή συζήτηση που είναι πιο απαραίτητη από ποτέ ενώπιον ε, της ε, ε, ανάδυσης των, ακροδεξιών δυνάμεων και στην Ισπανία. Ωστόσο, δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με τους, για την διάγνωσή σας με τις λύσεις που δίνεται σε όλους αυτούς τους κινδύνους που έχουν αναδεθεί. Σε σχέση με την ακροδεξιά, αυτά τα σχήματα φασιστικών τάσεων θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και να τις ε, κόψουμε από τη ρίζα. Αυτά τα φαινόμενα στην ουσία ε, οφείλονται στις ε, περικοπές που έχουν κάνει πολλές κυβερνήσεις ε, έναντι των εργατικών τάξεων. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν μειώσει στο σε πολύ μεγάλο βαθμό το κράτος πρόνοιας και η διαχείριση της κρίσης είναι και αυτή υπεύθυνη για μια αβάσταχτη ανισότητα. Με τις πολιτικές στην υπηρεσία των προνομιούχων έχετε προκαλέσει μια, ένα μεγάλο κοινωνικό ε, πόνο και μια κοινωνική κρίση και η Ισπανία συμμετείχε στις πικρές αυτές ε, στιγμές που ζούμε. Η συνταγματική μεταρρύθμιση εξπρέση και οι περικοπές στην παιδεία, στην υγεία, στις συντάξεις, ε, δύο εργατικές ε, μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα ζημιογόνες για τους εργαζόμενους. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτά όλα δημιούργησαν το, το, κατάλληλο λίπασμα, το κατάλληλο έδαφος ώστε η ακροδεξιά να εκμεταλλευτεί την απελπισία της κοινωνίας κοινωνικής και να παρουσιάσει ψευδείς εχθρούς και ψευδείς λύσεις. Ε, κύριε Σάντζες, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει πάνω από 140 εκατομμύρια φτωχούς και επισφαλείς εργαζόμενους. Συνέπεια και αυτό της ε, εδαφικής ασυμμετρίας του παραγωγικού μοντέλου μέσω του οποίου ζημιώνεται το, ο νότος της Ευρώπης. Μας καταδικάζουν σε υποβοηθούμενα μοντέλα που βασίζονται σε, χαμηλά αμοιβόμενα εργατικά χέρια. Θέσεις επασχόλησης που κρέμονται από, ένα, από μια κλωστή γιατί οι επιχειρήσεις ε, ε κοιτούν μόνο το κέρδος τους, ε, τα κέρδη τους. Αλκόα, Vodafone, Deliveroo, Amazon, ένα, ένας τεράστιος κατάλογος, δεν χρειάζεται να σας το διαβάσω όλα. Αυτά είναι το αποτέλεσμα όταν αφήνουμε τη δημοκρατία στα χέρια των πολυεθνικών, όταν η προτεραιότητα είναι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπου και αν βρίσκονται και από όπου και αν προέρχονται. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε δημόσιες πολιτικές που θα προωθούν τις ποιοτικέ θέσει απασχόλησης και θα εμποδίζουν ναι, την εργασιακή εκμετάλλευση σε οποιαδήποτε από τα κράτη-μέλη, γιατί μέχρι τώρα η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων έχει προχωρήσει παράλληλα με την ελεύθερη κυκλοφορία τη φτώχεια και τη ανισότητα. Οι οικονομικέ πολιτικέ ε, ε, ε, ε, της, δεξιάς μην τη συνεχίζεται, μην προβαίνετε σε στήρε ή συμμαχίες επιτεθείτε στα προβλήματα που επηρεάζουν τις, την εργατική τάξη. Δεν χρειαζόμαστε δεσμεύσει. Για παράδειγμα, ώστε η κοινωνική πολιτική να μετατραπεί σε ευρωπαϊκή πολιτική, να πιέζεται ώστε να επικυρωθεί ο ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη. Αυτό είναι ένα καλό κοινωνικό συμβόλαιο. Να κάνουμε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ένα παράγοντα σταθερότητα και όχι ε, και όχι αντιφάσεων όπως ας πούμε στην Δυτική Σαχάρα και στην Παλαιστίνη. Ε, ε, εκλογικός νόμος, ε, ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, απειλείται η δεξιά, την έχουμε οι γυναίκες, την έχουμε ζήσει στο πετσί μας, είναι διαρθωτική, θα συνεχίσουμε ωστόσο να αγωνιζόμαστε για να περασπιστούμε τα κοινά μας συμφέροντα των γυναικών. Ευχαριστώ. Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία, η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Πρόκειται για την 15η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης που γίνεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για 15η φορά πρέπει να επαναλάβουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια πολύ δύσκολη στιγμή και για 15η φορά πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο και η απάντησή μας είναι πάντοτε η ίδια. Λάθος πολιτικές, ε, αδικίες. Να σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Οι πολιτικές λιτότητες έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στην κοινωνία μας. Εχθές ο πρόεδρος Γιούνκερ παραδέχτηκε σε αυτή την ολομέλεια ότι, ότι αυτές οι πολιτικές λιτότητες κάποιες ζημιές έχουν κάνει. Καλό, καλή αργά παρά ποτέ λέμε, αλλά εδώ όχι, έχουμε ήδη ξεπεράσει τα όρια. Έχουμε δημιουργήσει οικονομίες που έχουν διαλύσει το σύστημα προστασίας των εργαζομένων και των πιο ευάλωτων κατηγοριών, αφήνοντας ε, ανικανοποιητές τις ανάγκες και ε, ε, δημιουργώντα ανθρώπου που δουν σε δυσκολία, δράμα τη φτώχεια, το δράμα τη έλλειψη απασχόληση και ο κοινωνικό αποκλεισμό που ζουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δεν σημαίνει ότι είμαστε λαϊκιστέ. Σημαίνει ότι διαπιστώνουμε την πραγματικότητα και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσει. Ο Γιούνκερ και άλλοι επίτροποι εκμεταλλεύονται του τελευταίου μήνε που του μένουν στην Κομισιόν για τι επόμενε εκλογέ θα υπάρξει αλλαγή μεγάλη, όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά σε ολόκληρη την Επιτροπή. Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να αναφέρω ως λανθασμένες πολιτικές έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές πολιτικές. Εδώ η αποτυχία της Ένωσης, μιας Ένωσης που είναι μόνο στα όνομα Ένωση και όχι στην πράξη, είναι προφανής. Η έλλειψη κοινή θέση για την ισότιμη κατανομή των ευθυνών και την αλληλεγγύη στις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη βήθησαν το μεταρρύθμιση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, όσον αφορά το άσυλο. Αυτό σημαίνει πως ε, οι περισσότερες τα περισσότερα προβλήματα βαραίνουν τα συνοριακά κράτη κυρίως και τους λιγοστούς συνεργάτες τους. η αποτυχία αυτών των ευρωπαϊκών πολιτικών έχει μεγάλο αντίκτυπο και μεγάλο κοινωνικό κόστος και οικονομικό κόστος που εκτιμάται στα 49 ε, δις ευρώ σύμφωνα με πρόσφατη ε, μελέτη. Δεν είναι η αλληλεγγύη μόνο που λείπει. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι δύο χώρε τη Μεσογείου που έχουν τα ε, παρόμοια συμφέροντα, όπω α πούμε για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την οικονομία. Όμω, βλέπουμε την έκφραση δύο διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων. Ωστόσο, οι χώρε μα θα πρέπει να συνεργαστούν για να καταπολεμήσουν τα προβλήματα και να βρουν λύσει για τα μεταναστευτικό. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συμβάλλει. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να δώσουμε και άλλα μηνύματα στους πολίτες. Οι πολίτες μας ζητούν συγκεκριμένες δράσεις και απαντήσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να περικόψουμε και τις ε, σπατάλες και ας ξεκινήσουμε από αυτήν εδώ, ε, αυτό εδώ το κοινοβούλιο, αυτή την άχρηστη και αδικαιολόγητη τριπλή έδρα. Ε, δισεκατομμύρια σπαταλώνται κάθε χρόνο για τα πήγαινέλα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να, να, να καταργηθεί αυτή η σπατάλη. Αυτό δεν σημαίνει κατάρριση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν είναι, δεν είναι προνόμιο, ούτε ένα κτίριο μόνο. Η λιτότητα, τις σπατάλες, οι πολίτες μας ζητούν αλλαγές. Θα πρέπει οι άνθρωποι να μπουν στο επίκεντρο των πολιτικών και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό τώρα τα δικαιώματα και η ευημερία όλων των πολιτών και να μην θυσιάζονται στο όνομα συγκεκριμένων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ε, συμφερόντων που ευνοούν μόνο λίγους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από ένα χρόνο βρεθήκατε τυχαία στο επικεφαλής της Ισπανίας χάρη λόγω του σκανδάλου που αντιμετώπισε ο Ραχώη. Ε, ωστόσο το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει μόνο 90 ε, έδρες. Είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα για την Ισπανία. Η πρώτη σας κίνηση ήταν να δεχτείτε το Aquarius. Ένα σκάφος το οποίο υποστηρίζει την παράνομη διακίνηση μεταναστών στην ε, Μεσόγειο, τη μαφία η οποία ε, πλουτίζει εκμεταλλευόμενοι τις ανθρώπινες ζωές. Οι διακινητές είναι αυτοί οι οποίοι υποφελούνται από την ε, διακίνηση αυτών των πλοίων όπου στηβάζουν τους μετανάστες. Ο Μακρόν και η Μέρκελ ε, ε, έσπευσαν να σας συγχαρούν. Ε, δεχθήκατε τις δύο, δύο φορές την κυρία Μέρκελ. Ε, χωρίς να διαβολευτείτε τους Ισπανούς, συνήψατε μία συμφωνία με την Καγκελάριο για να αντιμετωπίσετε το μεταναστευτικό. Ε, στο ζήλο σας ε, δεν συνειδητοποίησατε ότι ε, μιλή, αναφέρθηκε στο Μαρόκο μιλώντας για μια αβυσαλαία ανισότητα. Ε, αυτή όμως είναι η πιο ευημερούσα χώρα ε, στην περιοχή. Μια συμφωνία επανεισδοχής είναι, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη. οι πρόσφυγες βέβαια μετά από την πολιτική που εφαρμόσατε έσπευσαν στις πόρτα σας. Ε, στη Θέουτα και την ε, Μελίγια ε, προσπαθώντας να παραβιάσουν τα σύνορα καμιά φορά και με τη βία. Είσαστε υποτελεί στο Βερολίνο αλλά και στις Βρυξέλλες. Το 2011 η σοσιαλιστική ομάδα έσπευσε να προβεί σε μια μεταρρύθμιση του Ισπανικού Συντάγματος όπου ε, η κυβέρνηση ε, ε, δεσμεύεται να δεχτεί τα όσα της βάλλονται από την Κομισιόν. Ωστόσο, ο Ισπανικός λαός πλέον αφυπνίζεται. Δείτε τι έγινε στην Αδαλουσία ε, και αναφέρομαι στο συνασπισμό κυβέρνησης που έδιωξε από αυτό το προπήγιο του σοσιαλισμού τους, ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ε, το 2018 εξαιτία σας η αύξηση των μεταναστών αυξήθηκε, ήταν δραματική. Στην Ιταλία, ωστόσο, το ποσοστό αυτό έπεσε σημαντικά γιατί οι Ιταλοί απέστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ε, διακινητές. Ο Ματέο Σαλβίνη ε, δεν δέχεται ε, την εμπορία ανθρώπων η οποία αποφέρει περισσότερα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών. Κύριε Πρωθυπουργέ, η επίλυση του μεταναστευτικού είναι συνάρτηση πολιτικής ε, βίλησης, βούλησης, γιατί ε, οι δικές σας ε, υπηρεσίες ακτοφυλακής είναι εξίσου αποτελεσματικές με τις αντίστοιχες ιτηλικές. Αλλά αντί να στηριχθείτε σε αυτούς, κάνετε προσπάθειες, δημιουργείτε ταμεία για την καλύτερη ένταξη των μεταναστών. parola all'onorevole non iscritto. Ο και μη εγγεγραμμένος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη δουλειά του, για την ε, ομιλία του. Ο Πρωθυπουργό της Ισπανίας, όταν έρχεται εδώ πέρα, δεν εκπροσωπεί το πολιτικό του κόμμα, αλλά εκπροσωπεί κυρίως τη χώρα του. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανία για όλες τις προσπάθειες της μέχρι στιγμής. Ακούσαμε τον συνάδελφο Φερχόφστατ που μίλησε για τον φεντεραλισμό. Η Ευρώπη σήμερα χρειάζεται πιο πρακτική προσέγγιση, περισσότερο σεβασμό για τις χώρες, ανταγωνιστικότητα ε, στην οικονομία και λιγότερο συγκεντρωτισμό. Αυτά ήθελα να ακούσω. Επίσης φαίνεται ότι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με την αλληλεγγύη αλληλεγγύη είναι όταν βλέπω να υπάρχει ανάγκη να βοηθήσω κάποιον άλλον. Όταν κάποιος ε, έχει βρεθεί σε ατυχή θέση χωρίς ε, να ευθύνεται ο ίδιος. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πληρώνω για την ανευθυνότητα των άλλων. Η Ισπανία θα είναι σημαντικός μας εταίρος κατά τη συζήτηση μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο ο κύριος ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους παρεμβαίνοντας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό τον γύρο συζήτησης. Αν μου επιτρέπετε, ε, ε, θα ήθελα να πατήσω στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων από κοινού, όχι στον καθένα προσωπικά, γιατί αυτό θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Η κεντρική ιδέα τη παρέμβασή μου είναι ότι θα πρέπει να προστατευτεί η Ευρώπη, ούτω ώστε η Ευρώπη να μα προστατεύσει και αυτή. Και πολλέ από τι παρεμβάσει των πολιτικών ομάδων έδειξαν ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη, ε, γευρώνοντα τι ε, πολιτικέ μα διαφορέ. Το ερώτημα είναι σε ποια κατεύθυνση. Και θα ήθελα να αναφερθώ πρωτίστω στο θέμα τη μετανάστευση. Ε, Βεβαίω ε, ισχύει τα ε, ε, δεν ισχύει το ότι η μετανάστευση ε, έφτασε μαζί με, το, με την άνοδο των σοσιαλιστών στην εξουσία. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι η μεταναστευτική πολιτική στην Ισπανία, η οποία στο παρελθόν δεν είχε απολύτως κανένα νόημα. Εμείς πάντοτε ε, γνωρίσαμε τι γίνεται και αποφασίσαμε να δεχτούμε το Aquarius, γιατί γνωρίσαμε ότι η πρόκληση τη μετανάστευση απαιτεί από όλε τι χώρες, από όλε τις χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κοινή ε, θέση πρωτίστω το ανάληψη ευθύνη και δεύτερον την αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση τη Ισπανία ε, έχει μια εξωτερική ε, πολιτική όπω αυτή η οποία ανέπτυξε ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωσης. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν βάσει των κονδυλίων να ενισχύσουμε την Αφρική. Εμείς εδώ ε, και μήνες έχουμε διμερείς ε, διαλόγους με το Μαρόκο και όλες τις χώρες του Σαχέλ, όχι μόνο ε, για τα συμφέροντα να προσπίσουμε τα συμφέροντα της Ισπανίας, αλλά και ολοκλήρου της Ευρώπης. Η Ισπανία εδώ και πολλά χρόνια έχει μια πολιτική επιστροφής με το Μαρόκο, τη Μαυριτανία και άλλες χώρες της περιοχής. Εγώ πήγα στο Μαλί, όπου προσπαθήσαμε να, να επανεκκινήσουμε μια πολιτική εκούση ε, επιστροφής των υπηκών του Μαλή που αυτή τη στιγμή ζουν στην Ισπανία. Ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε λοιπόν αυτή την πολιτική επιστροφής ε, και προσπαθούμε επίσης να ενισχύσουμε την πολιτική στα σύνορα. Και χωρίς αμφιβολία αυτό που κάνουμε να ενισχύσουμε ε, την πολιτική ένταξη. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε αυτή την πολιτική ένταξη για όλους τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και χωρίς αμφιβολία θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε υπέρ μιας μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χορήγησης Ασύλου. Ε, εμένα, εγώ εδώ έχω πολλές ανησυχίες όσον αφορά το Σέγγεν, γιατί υπάρχουν πολιτικές ομάδες όπως το ΕΛΚ που δεν συνεργάζονται εδώ. Με ανησυχεί λοιπόν η κατάσταση αυτή. Εμένα δεν με ανησυχεί τόσο πολύ η παρουσία της ακροδεξιάς. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι το πώς η ακροδεξιά παρισφρεί στην ατζέντα ε, πολιτικών κομμάτων που υποτίθεται ότι ήταν ε, φιλοευρωπαϊκά. Ε, η κυβέρνηση αυτή, κύριε Φερχοφσάτ, στηρίζει χωρίς αμφιβολία την έγκριση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, το υπερασπιστήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την ε, προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Ραχώη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εγκριθεί πριν από τις ευρωεκλογέ γιατί είναι θεμελιώδες για την ε, γεωργική πολιτική στην Ισπανία, πολιτική συνοχή και άλλες σημαντικές πολιτικές όπως είναι η πολιτική μετανάστευσης ή πολιτικές που συνδέονται με ζητήματα καινοτομίας εμείς ε, θα εγκρίνουμε τον ε, προϋπολογισμό της χώρας κατά πάσα πιθανότητα τον Απρίλιο. Ε, άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται να προβούμε στην έγκριση του προϋπολογισμού γιατί θεωρούμε ότι είναι θετικός όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την αναδιανεμετική πολιτική και περιλαμβάνει καινοτομίες όσον αφορά το φορολογικό σύστημα, για παράδειγμα η δημιουργία φόρου επί των συναλλαγών και αυτά είναι κάποια από τα μέτρα που εσείς οι ίδιοι προτείνατε σε αυτό το σώμα και εμείς προωθούμε στο επίπεδο της εθνικής μας πολιτικής. Ε, επιτρέψατε μου επίσης να αναφερθώ για την Καταλωνία, γιατί ε, το έκανε η ε, επικεφαλής της πολιτικής ομάδας των Πρασίνων. Από το 2014 έγιναν πέντε ψηφοφορίες, ε, τρεις εκλογικές διαδικασίες σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των δημοψηφισμάτων και αυτών των εκλογών ε, στο πλαίσιο του συνταγματικού ε, του Ισπανικού Συντάγματος. το 62% δεν υπερψήφισε την απόσχηση. Οι αποσχεστικές τάσεις δεν έχουν κοινωνική πλειοψηφία. Το 52% στην Ισπανία δεν είναι υπέρ της ε, απόσχησης. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να επιβληθεί ένα πολιτικό σχέδιο σε μια πλειοψηφία η οποία δεν συμμερίζεται την ε, απόσχηση. Πρώτο λόγο πρώτος λόγος είναι αυτός. Δεύτερον, είναι προφανές ότι στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Καταλωνία, εάν δούμε τι γίνεται για παράδειγμα στη Βαυαρία ή εάν δούμε τι γίνεται στο Βένετο στην Ιταλία ή στη Γαλλία, στην Κορσική, υπάρχουν εδαφικές ε, τάσεις, υπάρχουν ε, κινήματα εδαφικής ε, διάσπασης. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτό που συνέβη στην Καταλωνία και αυτό που συνέβη στο Βένετο ή για παράδειγμα στην ε, Βαβαρία όταν διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί ήθελαν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία της Βαβαρίας ή του Βένετο στην Ιταλία. Ή όταν το Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δικαστήριο του Βένετο στην Ιταλία ή ε, ε, αυτό που έγινε στη Βαβαρία. Στην ε, Ισπανία υπήρξαν κατ' επανάληψη αποφάσεις ε, του δικαστηρίου όπου υπόθηκε ότι δεν είναι δυνατή η απόσχηση. Ωστόσο, δεν εκπληρώθηκε αυτή η εντολή εκ μέρους των περιφερειών που επιθυμούν την απόσχηση. Από το 2010 η Καταλωνία έχει ένα σύνταγμα το οποίο στο σύνολό του δεν υπερψηφίστηκε από τους ε, πολίτες. Εδώ και δέκα χρόνια είναι προφανές ότι τα πολιτικά κόμματα όταν είναι στην αντιπολίτευση ε, χρησιμοποιούν ε, το θέμα της Καταλωνίας για να πιέσουν την κυβέρνηση. Ε, εμείς θα ακολουθήσουμε την πολιτική μας. Η Ισπανία είναι μια σημαντική χώρα η οποία έχει ένα υψηλό επίπεδο αποκέντρωσης, όχι μόνο οικονομικής αλλά και και πολιτιστική όσον αφορά την αναγνώριση των διαφορών γλωσσών και όσον αφορά τα παιδιά ε, που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ένα εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ε, εθνικό, ε, διαφορετικής, που έχουν διαφορετική εθνική προέλευση. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι προφανές ότι στην Καταλωνία θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινής ε, διάλογος και να αναγνωρίσουμε ότι στην ε, Καταλωνία η πλειοψηφία δεν είναι εθνικιστική. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν ένας διάλογος μεταξύ εθνικής κυβέρνησης και Καταλωνίας όσον αφορά την εθνικιστική, το εθνικιστικό και μη εθνικιστικό κομμάτι στην ε, Καταλωνία. Και βεβαίως ε, σημαντικό είναι το να έχει η ισπανική κυβέρνηση την πολιτική βούληση να επιλύσει το ζήτημα της Καταλωνίας. Αλλά θα πρέπει όπως είπα να αναγνωρίσουμε ότι οι αποσχετικές τάσεις δεν έχουν την πλειοψηφία στην Καταλωνία. Και ε, θέλει η κοινωνία της Καταλωνίας επιθυμεί μία λύση για, να, για το πρόβλημα αυτό. Η λύση που θεωρώ ότι υπάρχει στο ζήτημα των μεσογειακών τάσεων είναι η βούληση να υπάρξει δυνατότητα συνύπαρξης. Τέλος, ο κ. Βέμπερ έκανε μια αναφορά στην πρόταση Μομφής. Η πρόταση Μομφής είχε μια εντολή δηλαδή η δημοκρατική αναγέννηση της χώρας μας. Αυτό που συνέβη στην Ανδαλουσία, ανάμεσα στο ε, Λαϊκό Κόμμα, τους φιλελεύθερους και τους ε, αδερφούς του, ε, του Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας, είναι μία ε, συνεργασία των δικαιωμάτων, μια συγχώνευση των δικαιωμάτων, όπως ας πούμε για την ισότητα των φίλων και την καταπολέμηση της ε, έμφυλης βίας. Στην Ανδαλουσία λοιπόν πέρασε, πέρασε ένα σύνορο το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κάνει συμμαχία με την άκρα δεξιά. Ποτέ δεν πρόκειται εμείς να το κάνουμε αυτό ε, όπως κάποιοι είπαν με τις θέσεις τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να σας πω ότι η θέση της Ισπανικής κυβέρνησης είναι υπέρ της Ευρώπης. Αυτές είναι οι προτάσεις που είχαμε να κάνουμε. Τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, τη στρατηγική ή μάλλον καλύτερα την καταπολέμηση της επισφάλειας στην εργασία, την ε, ανεργία των νέων, ε, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της Ευρώπης ώστε να μας προστατεύσει καλύτερα, ιδιαίτερα να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους, σίγουρα στην, Ευρωπαϊκή, στην Ισπανική κυβέρνηση και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα θα βρουν σύμμαχο. Κύριε Φερχόφσας, να σας πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε πως... Ε, Εσεί είστε πολλά χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και εγώ μόλι 7 μήνε στην κυβέρνηση τη Ισπανία και σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε τα προβλήματά μα. Όμω, πιστεύω πω θα πρέπει να βρούμε και εξόδους αυτό το, την έλλειψη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων που χρειάζονται στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εξωτερική Πολιτική. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αλλαγή των διαδικασιών λήψη απόφαση στο Συμβούλιο και στο, στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Και σίγουρα, όπω το είπα ήδη, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουν ε, οι κανόνες ώστε να μην λαμβάνονται αποφάσεις ομόφωνα μόνο. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, θα χρειαστεί βέβαια αλλαγή στις συνθήκες, για άλλα πράγματα όχι. Ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μπορέλ, μόλι μου θύμωσε, θύμισε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι πασαρέλε που υπάρχουν ε, στι συνθήκε για να ενισχύσουμε τον γενικό χαρακτήρα της Υπήρου μας ε, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάμε με το Catch the Eye. Καθυστερούμε λίγο τις ψηφοφορίες σας. Παρακαλώ να σεβαστείτε το ένα λεπτό, γιατί όσο περισσότερο το σεβαστείτε, τόσο περισσότερο θα πάρετε και το λόγο. 150 έχουν ζητήσει το λόγο. Πόνς. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή ψευδών ειδήσεων, αλλά επίσης και όπως είδαμε και σε μια εποχή ε, σφαλμένων και ψευδών επεπιθύσεων. Με, το, με την ψήφο των, ε, πρώην τρομοκρατών και της άκρο αριστεράς βρίσκονται στην εξουσία. Η αυτή η κυβέρνηση. Και μόνο με τις ψήφους των αποσχιστών, των πρώην τρομοκρατών και της ακροαριστεράς θα μπορούσαν να σταθούν. Οι πρώτη σας ομιλίες μιλήσατε πολύ για την παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν μπορέσατε να μιλήσετε για την ενότητα της Ισπανίας και δεν μπορέσατε να υπερασπιστείτε το κράτος δικαίου. Μιλήσα, θα σας πω κάτι για την Καταλωνία. Αυτό που είπατε είναι, είναι ότι δεν είναι πρόβλημα ανεξαρτησίας, αλλά πρόβλημα συμβίωσης. Ενώ το ανώτατο δικαστήριο α, ξεκινά τέτοια διαδικασία και όλοι περιμέναμε τον πρόεδρο της Ισπανικής κυβέρνησης να υπερασπιστεί το κράτος δικαίου της χώρας μας. Και το λέω ως Ισπανός βουλευτής. Δύο χρόνια υπερασπιζόμαστε και τους δικούς σας βουλευτές εδώ για την ενότητα της Ισπανία, Αλλά το να υπερασπιστείτε την ενότητα της Ισπανίας δεν είναι μόνο θέμα της θέσης σας, αλλά είναι και θέμα πεποίθησης, πε, πεποίθησης που να μην είναι ψευδής. Δυστυχώς, επειδή είστε πρόεδρος της Ισπανίας στην στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν σας βγήκε εσείς, εσ, εσείς δυστυχώς δεν μπορέσατε να το κάνετε. Με, με αλλά κάνω υπομονή. Κυρία Γκαρσία Πέρες, Πρόεδρε Σάντσες. Είναι ευαίσθητη, λεπτή στιγμή για την Ευρώπη. Και το να ακούμε την ομιλία σας με δέσμευση σαφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ανανάσα για όσους πιστεύουμε ότι η λύση στα προβλήματά μας βρίσκεται στην Ευρώπη, σε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντισταθούμε στον πειρασμό να φέρουμε αυτά τα επιχειρήματα στη Μαδρίτη για να κερδίσουμε, να, να μην διστάσετε μάλλον να τα φέρετε στη Μαδρίτη για να κερδίσετε πόντους. Αλλά δεν θα εξυπηρετήσουμε την Ευρώπη αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο και την καρδιά της Ευρώπης για να μιλήσουμε για το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερη ισορροπία, να αποφύγουμε τις ανισότητες, να προωθήσουμε μια Ευρώπη όπου να υπάρχει ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, να μπορούμε να κοιτάξουμε στο καταπρόσωπο τους, τους πολίτες και να πούμε πως η Ευρώπη είναι τη λύση για τα προβλήματα. Αυτή είναι η δέσμευση των Ευρωπαϊστών, της σοσιαλδημοκρατίας και θα πρέπει να, να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια ώστε να περισπιστούμε περισσότερη Ευρώπη που θα μπορεί, όπως είπα, να κοιτάξει κατά πρόσωπο τους πολίτες. Και ευχαριστώ πολύ που μπορείτε να έχουμε να έχουμε κυβερνήσεις ε, μέσα στην Ευρώπη που, θα που εξακολουθούν να στηρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Η πολιτική ξεκινάει με την παρατήρηση της πραγματικότητας, έχει πει ένας ε, γνωστός ε, σοσιαλδημοκράτης ε, και γι' αυτό γιορτάσαμε την επέτειο του ευρώ και άκουσα έξι ομιλίες που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλλον επιθυμίες εξέφραζαν. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλετε κοινωνική Ευρώπη. Η κοινωνική Ευρώπη δίνει δουλειά στους ε, πολίτες και προοπτικές στους νέους. Αυτό είναι αποφασιστική σημασίας. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία στους νέους, ε, γιατί δεν ε, έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις, ε, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στην Ευρώπη. Υπάρχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες. Εργαζόμαστε όλο και περισσότερο για λιγότερα χρήματα και δεν είναι αυτή η κοινωνική Ευρώπη που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αντιμετωπίζουμε την απειλή των λαϊκιστών και αποσχιστών. Αλλά δεν αρκεί η καταγγελία. Θα πρέπει να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις στην αιτία που είναι η αλλαγή μοντέλου η σύγχυση που επικρατεί στην οικονομία. Ωστόσο σήμερα όλα έχουμε δόγματα παρά λύσεις. Κύριε Σάντσεθ, η λύση δεν είναι με τους λαϊκιστές της αριστεράς ή της δεξιάς που θέλουν να αποδυναμώσουν την Ευρώπη ενώπιον του λαϊκισμού και της απόσχεσης των αποσχιστικών τάσεων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδημήσουμε την Ευρώπη και να την υπερασπιστούμε. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω σε εκείνους που θεωρούν ότι η Καταλωνία είναι πρόβλημα των Καταλανών, ότι στην Καταλωνία το πρώτο κόμμα το οποίο αναπτύσσεται στην Ισπανία είναι το κόμμα Σιουδαδάνος, όχι κόμμα αυτονομιστών. Αρκεί τον, φτάνει, δεν χρειάζεται να προβάλλουμε άλλα συνθήματα. Ε, βασική μας αρχή θα πρέπει να είναι η ελεγγύη και η ενότητα. Αυτό ισχύει τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ισπανία. Κύριε πρόεδρε της Ισπανικής Κυβέρνησης. Στις 5 Νοεμβρίου του περασμένου έτους ε, πήγα να επισκεφτώ τους παλιούς συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σήμερα είναι φυλακισμένοι στις Ισπανικές φυλακές. Ε, κάτι που σήμερα ε, είναι αδιανόητο να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Άνθρωποι οι οποίοι εξελέγησαν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια στην Καταλωνία με νόμιμο τρόπο να φλαγίζονται για τις ε, πολιτικές τους ιδέες. Έχουμε στο Κοινοβούλιο αυτό κατ' επανάληψη πει και καταγγείλει τις ανελεύθερες ε, πολιτικές του κυρίου Ορμπάν. Έχουμε καταγγείλει την ανελεύθερη πολιτική της Πολωνίας. Έχουμε καταγγείλει απολύτως δικαιολογημένα τις επιθέσεις στα δικαιώματα που σήμερα λαμβάνουν χώρα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν η Ισπανία λόγω ακριβώς του συντάγματός της και της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται στην Καταλωνία προσχωρεί στο στρατόπεδο αυτών των χωρών. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι κρίμα. Άκουσα την ομιλία σας. Αλλά πώς είναι δυνατόν ε, σήμερα ε, άτομα βουλευτές συγκεκριμένα μέλη περιφερειακών κυβερνήσεων και ε, ενώσαν να είναι φυλακισμένοι. Άκουσα την έκκλησή σας ε, για το διάλογο και τη συμμερίζομαι αλλά θα πρέπει να απελευθερώσετε άμεσα αυτά τα άτομα προκειμένου να υπάρξει διάλογος. Ε, θα πρέπει να αναλάβετε τις ε, ευθύνε σας. Ε, απελευθερώστε άμεσα τα άτομα αυτά, μόνο έτσι θα αποδείξετε το δημοκρατικό σας πνεύμα. Ε, Πρώτα σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε το σύστημα DONT. Εάν δεν τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης, ε, αυτό θα είναι σε βάρος ενός συναδέλφου. Αυτό είναι ο κανόνας και θα πρέπει να την, ε, το σεβαστεί το κύριο Σορμπαν Κρέσπο. Κύριε Σάντσες, η κυβέρνησή σας ξεκίνησε υποδεχόμενη το Aquarius και έξι μήνες αργότερα τελείωσε μπλοκάροντας το Open Arms στη Βαρκελόνη και σίγουρα προς χαρά φασιστών όπως ο Σαλβίνη. Υποσχεθήκατε την εξαίρεση ε, και την άρση του νόμου Φήμοτρο, αλλά συνεχίζει να ισχύει. Υποσχεθήκατε την ε, εργασιακή μεταρρύθμιση. Όχι μόνο δεν το κάνατε, αλλά επιτρέψετε και σε εταιρείε όπως η Αλκοα να απολύουν ε, εκατοντάδες εργαζόμενους. Υποσχεθήκατε φόρο στις τράπεζες, αλλά δεν έχει φτάσει. Υποσχεθήκατε να ρυθμίσετε τη φούσκα των μισθωμάτων που Διώχνουν από τα σπίτια τους εκατοντάδες ανθρώπους, αλλά τίποτα δεν κάνατε. Τελικά κερδίζουν ε, τα αρπακτικά νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε αυτές είστε ένοχοι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ε, μεγάλης συμμαχίας και στην Ανδαλουσία χρειαζόμαστε ε, μια στροφή 180 μοιρών από τις πολιτικές περικοπών που εξυπηρετούν τις ελίτ. Είναι σημαντικό να γίνει αλλαγή στην Ευρώπη. Δεν έχουμε πια χρόνο κύριε Σάντσε. Πρέπει να γίνει τώρα η αλλαγή. Ο κύριος Ντάρμος. Ε, Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Μπόβε σχετικά με τους Καταλανούς φυλακισμένους ε, που επί ένα χρόνο κρατώνταν πριν τη δίκη τους. Πρόκειται για πολιτικούς κρατούμενους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν κάνει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο δεν λέει τίποτα. Και ακόμη και ο κύριος Φερχόφστατ σιωπά. Οι ευρωπαϊκές αξίες για τις οποίες ακούμε συνέχεια ε, δεν γίνονται σεβαστές και αναρωτιέται κανείς γιατί η, η Ισπανική κυβέρνηση στηρίζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και γι' αυτό φαίνεται ότι είναι εντάξει το να έχει κανείς πολιτικούς κρατούμενους. Αυτό είναι λυπηρό. Η υποκρισία είναι πολύ δύσκολο να παταχθεί και καλό όλους σας να κοιταχτείτε στον καθρέφτη και να αρχίσετε εκστρατεία για απελευθέρωση αυτών των πολιτικών κρατούμενων. Ο κύριος Καλώ ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα να σας ε, υποβάλω. Ποια πρακτικά, σε, ποιε πρακτικέ ποιες πρακτικές ενέργειες θα προβείτε ούτως ώστε η χώρα σας, η Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η πατρίδα μου η Ελλάδα να πάψουν να είναι τόποι μόνιμης διαμονής παρανόμων μεταναστών. Είπατε ότι είστε υπέρ της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού στρατού. Για να δικαιολογείται όμως η αύξηση των δυνατοτήτων των στρατιωτικών τη ευρωπαϊκή ενώσεω θα πρέπει να υπάρχει ένα εχθρό ο οποίο θα απειλεί την ευρώπη. μπορείτε να μα κατονομάσετε ποιο είναι αυτό ο εχθρό και ποιε χώρε απειλεί διότι όπω ξέρετε και όπω γνωρίζω και εγώ οι μόνε χώρε τη ευρώπη που απειλούνται από τρίτη χώρα είναι η ελλάδα και η Κύπρο που απειλούνται από την τουρκία. είπατε επίση ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει έξω από τα σύνορά τη. αυτή είναι η ευρώπη του μέλλοντο που οραματίζεστε. ο ρόλο ενό παγκόσμιου χωροφύλακα υποστηρίξατε επίσης ότι πρέπει να καταργηθεί η αρχή της ομοφωνίας. όμως εάν καταργηθεί η αρχή αυτή τότε θα μειωθεί η δύναμη των κρατών και κυρίως των μικρών κρατών. μπορείτε να φανταστείτε τη χώρα σας να θίγεται να θίγονται τα συμφέροντά της να βρίσκεται στην θέση της μειοψηφίας και να μην μπορεί να υπερασπιστεί αυτά τα συμφέροντά της. ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Καταρχάς για μια πολύ επικοδομητική ομιλία. Είναι σαφές ότι ε, η Ισπανία είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης και η Ευρώπη είναι αξιόπιστος εταίρος της Ισπανίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, την πολιτική συνοχή σε την εγγύηση για τους νέους. Ας είμαστε σαφείς όμως, η ευθύνη για μια κοινωνική Ευρώπη ξεκινάει στα σπίτια μας, ε, στις πατρίδες μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι επικίνδυνη στρατηγική ε, να ε, ρίχνετε στην Ευρώπη το φταίξιμο για αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς ε, στη χώρα σας. Η Ισπανία βρίσκεται σε καλή θέση λόγω της καλής δουλειάς προηγούμενων κυβερνήσεων. Να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την εργασία και ας μην ρίξουμε σε επόμενες γενιές τον φόρτο. Η προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με την Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Κύριε Σήμερα εδώ μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης και δεν κατάλαβα γιατί τελικά η ομιλία σας ε, μετατράπηκε σε μια μικρή προεκλογική ομιλία υπέρ του κυρίου Τίπερμανς, Τίμερμανς. Και επίσης αναρωτιέμαι γιατί αυτοί που χρησιμοποιούν τους ε, παλιούς δικτάτορες για να καταδικάσουν άλλους γιατί δεν μιλάτε για τους σημερινούς δικτάτορες όπως της Βενεζουέλας και τις Κούβας. Εσείς θα ζητήσετε ε, κυρώσεις εναντίον αυτών των δύο ή θα συνεχίσετε μόνο με λόγια. Θα δείξετε αυτόν τον φιλοευρωπαϊσμό σας καταγγέλλοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μη στηρίζοντα τα δεκτατορικά καθεστώτα του Μπαντούρου και του Κάστρο γιατί ο Κάστρο είναι που ε, που ηγείται της Κούβας. Ε, υπάρχουν ε, πολιτικοί κρατούμενοι στην Κούβα και στη Βενεζουέλα και τότε θα πούμε και εμείς ότι είστε ευρωπαϊστής. Μπλάνκο Λόπεθ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Στέμπαν Γκοσάλε Πόνσε, το να είναι κανεί πατριώτη ε, δεν σημαίνει το να στηρίζει την Ισπανία, αλλά να τηρεί τις συνταγματικές και ευρωπαϊκές αρχές και όχι να ε, πάει χέρι-χέρι με αυτόν που θέλει να τις καταστρέψει. Εσείς είχατε την ευκαιρία να δείξετε ότι είστε πατριώτης ισπανό, Ισπανός, στηρίζοντας την κυβέρνηση της Ισπανίας, όπως ανέκαθεν κάναμε εμείς οι σιωλισσαλιστές, όταν η Ισπανία απειλεί το και εσείς ερχόσασταν να μας ζητήσετε βοήθεια. Εσείς όμως στάσατε στην κυβέρνηση τη Ισπανίας φωνάζοντας θα διαλυθεί η Ισπανία. Ενώ τούτη η Ισπανία ε, έλαβε μια Ισπανία, με κληρονόμησε μια Ισπανία πιο διχασμένη από ποτέ με συνύπαρξη και συμβίωση ε, χειρότερη από ποτέ. Δυστυχώς εσείς δεν συμβάλλετε στο να δημιουργηθούν χώροι συμβίωσης που είναι ακριβώς αυτό το οποίο στηρίζει η κυβέρνηση της Ισπανίας η σημερινή. Και ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμασιτς gospodine σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση αυτή. Μετά το δημοψήφισμα για το Brexit και με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ ε, κινούμαστε προς ε, μια πολύ κακή κατεύθυνση. Εσείς αναφερθήκατε σε σημαντικές προκλήσεις που δεν ε, σχετίζονται με την πολιτική ολοκλήρωση όπως είναι τα εργασιακά δικαιώματα και θέματα της κοινωνικής Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να είναι προπίδιο των ε, εργασιακών δικαιωμάτων για να είμαστε όμως ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα πρέπει να εισάγουμε αδικαιολόγητα υψηλούς φόρους και ε, αυστηρή, υπερβολικά αυστηρή νομοθεσία. Το θέμα αυτό σχετίζεται και με τις δημόσιες δαπάνες. Επί πολύ καιρό η Ισπανία αντιμετώπιζε προβλήματα. Ε, θα είναι σημαντική όμως για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, ε, αναμένουμε να ε, φέρετε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο να οικοδομείται με εμπιστοσύνη. Ε, εμείς η χώρα των Βάσκων θέλουμε να συμβάλλουμε στη σταθερότητα, να συμβάλλουμε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, ενισχύει το σύστημα κοινωνικής προστασίας, ε, προωθεί εγχειρήματα τα οποία επιφέρουν ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ενώπιον σύνθετων προβλημάτων χαιρετίζουμε τη βούλησή σας να τα επιλύσετε. Ε, ωστόσο, πουλάτε, δεν θέλουμε να πουλήσετε εσφαλμένες ε, συνταγές. Ε, θέλουμε να υπάρξει ένα μοντέλο συνύπαρξης, το οποίο όμως να εδράζεται στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί ένα πολιτικό πρόβλημα σε μια νομική υπόθεση. Ε, θα πρέπει να υπολογίστε στη δική μας ε, συνεργασία εάν ε, θέλετε να επιφέρετε αποτελέσματα χρήσιμα και υποφελή για τη συνύπαρξη, την ελληνική συνύπαρξη όλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σάντσεθ, χαιρετίζουμε την παρουσίαση του προπολογισμού στην Ισπανία γιατί ε, μας υπενθυμίζετε ότι είναι δυνατόν στην Ευρώπη ένας πιο σοσιαλιστικός κοινωνικός ε, δρόμος. Ε, απέναντι στην Ευρώπη του μίσους υπάρχει και το μοντέλο της βιώσιμης Ευρώπης. ένα μοντέλο πιο φιλόδοξο όσον αφορά την επίδειξη τόλμης έναντι του μεταναστευτικού ε, εφόσον επιτρέπεται την υποδοχή σκαφών που σώζουν ζωές και βαίνουμε προς, μια, ε, προς τη μετάβαση ενός πιο οικολογικού μοντέλου. Ε, είστε υπέρ των καθαρών συνεργειών, υπέρ της κλιματικής προστασίας, υπέρ της μείωσης των, της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια σας. Θα σας στηρίξουμε. Ο κύριος Κόμη. Καλημέρα σα, ε, Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσεί μιλήσατε πολύ για τι γυναίκε, για τα δικαιώματα των γυναικών, τη βία κατά των γυναικών. Εύχομαι την επόμενη φορά να μπορέσετε να μα έρθετε με κάπω πιο θηλυκό επιτελείο, γιατί σήμερα μόνο άνδρες βλέπω. Από τα λόγια να περάσουμε στι πράξει. Ε, ε, αυτή είναι η ευχή μου λοιπόν. Τώρα επειδή η Ιταλία και η Ισπανία ανέκαθεν ναι, είχαν καλή σχέση και, και για την μετανάστευση πιστεύω πως ε, εκεί μπορούμε να είμαστε οι εκπρόσωποι των χωρών της, Μεσογείου για τη μεταρρύθμιση της, μεταρρύθμιση της του Δουβλίνου. Και γιατί όταν λέμε ότι πως η Ευρώπη μας έφυσε μόνος, ε, υπάρχει όνομα και επίθετο. Είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν τα κράτη-μέλη. Το Ευρωκοινοβούλιο υπορψήφισε τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και τις ε, ε, μεταναστευτικέ ζωέ. Όμω εσεί και οι άλλοι πρωθυπουργοί θα πρέπει να συμφωνήσετε για το θέμα για τι κατά των γυναικών. Εμεί στο ΕΛΚΑ είμαστε υπέρ να υπάρξει ένας απολογισμός, ένας ε, σύνδεσμος που μπορεί να είναι αυτός των, ε, της απασχόλησης και της ε, οικογένειας και οι γυναίκες να μπορούν να εργάζονται και να μην κάνουν μόνο τις νοικοκυρές υποχρεωτικά και όχι από επιλογή. Ο κύριος Φέρμπερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ όταν συγκρίνεται την Καταλωνία και τη Βαβαρία. Θα ήθελα να ε, δίδεται ακριβή στοιχεία. Ε, πριν από 100 χρόνια υπήρξε μια ακροαριστερή ε, κίνηση για απελευθέρωση σε μια εποχή που δεν υπήρχε το βασίλειο της Γερμανίας. δεν είναι συγκρίσιμη με την περίπτωση της Καταλωνίας η περίπτωση αυτή. Δεύτερον, ε, είπατε τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τι κάνει η κυβέρνησή σας. Ε, δεν αρκεί να απαιτείτε λύση στην ανεργία από πλευρά της Ευρώπης ε, τη στιγμή που ανακαλείτε ρυθμίσει της προηγούμενης κυβέρνησης για απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Εσείς δηλαδή δεν λαμβάνετε μέτρα για την απασχόληση των νέων. Ε, ήθελα να ακούσω περισσότερα για το θέμα αυτό. Δεν αρκεί να ζητάτε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα πρέπει κανείς να λαμβάνει και μόνος του μέτρα. Ε, είναι θέματα αλληλένδετα ε, μεταξύ τους αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ. Köszönöm a Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε εδώ για το μέλλον της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχουν ε, κυβερνήσεις κρατών μελών ε, που ε, δεν δέχονται ανθρώπινα δικαιώματα και δημιουργούν ένα σύστημα μη ε, φιλελεύθερο και αναφέρομαι στην Ουγγαρία και ε, τον Βίκτορ Ορμπάν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, έχουν αλλάξει και οι βουλευτές δεν κάνουν τίποτα. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αποκτήσει τεράστιες περιουσίες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών πεινούν. Επίσης ε, παρενοχλούνται ε, άνθρωποι ε, της κοινωνίας των πολιτών. Η Ισπανία από δικτατορία έχει γίνει μια σεβαστή δημοκρατική χώρα. Τι πρέπει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε τις δικτατορίες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Αν μιλάτε το διπλάσιο από το χρόνο που σας έχει δοθεί, παίρνετε το χρόνο των συναδέλφων σας. Στη μία η ώρα θα ψηφίσουμε. Καλωσορίσατε ορίσατε κύριε Σάντσε, ε, κύριε Δεμεσμάκερ. Στις 21 ε, Δεκεμβρίου ήμουν στη Βαρκελόνη και εσείς ήσασταν εκεί. Ε, Τέσσερι Καταλανοί κρατούμενοι είχαν μόλις σταματήσει την απεργία πείνας. Εγώ δεν ε, μου πέφτει λόγος για τις πολιτικές σας και τις στρατηγικές σας. Αυτό που δεν δέχομαι όμως είναι ότι ο κόσμος τώρα εδώ και πάνω από χρόνο βρίσκεται στη φυλακή λόγω και κατηγορούνται για ε, απόσχηση. Κανένας δεν έχει κάνει ε, βίαιη ε, επανάσταση και δεν το βλέπουμε αυτό σε ε, χώρες όπως η δική μου. Οι πολιτικές επιδιώξεις στηρίζονται μέσω του, διαλόγου νομίζω πως έχετε χάσει εδώ εν, μια στιγμή. Υπάρχει, υπάρχει επικίνδυνη νοσεθνικισμός στην Καταλωνία, ε, όχι όμως στην Καταλωνία με συγχωρείτε, αλλά ε, αλλού όπου αναβιώνει ο φραγκισμός και ελπίζω πως θα ξεπεράσετε το φόβο σας ε, των άκρων και θα απελευθερώσετε τους πολιτικούς κρατούμενους. Ο κύριος Τρεμόζα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Σάντσε, Κύριε Μπορέλ, καλώ ήρθατε και πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, δημιουργήθηκε ένα φοβερό προηγούμενο